the switching off. E, proszę Państwa, Panie i Panowie, proszę o zajęcie miejsc na sali. Rozpoczynamy posiedzenie. Παρακαλώ καθίστε, θα ξεκινήσουμε την συνεδρία της Ολομέλειας. Κυρίσω την έναρξη της Ολομέλειας που διακόπτει την ε, 20 Μαρτίου 2010. Πρώτα απ' όλα τα ανακοινοθέντα. Οι ανακοινώσεις μάλλον πριν από μερικές μέρες ε, πολλά άτομα στην Μόσχα έχασαν τη ζωή τους μετά από μια τρομοκρατική ενέργεια στον ε, υπόγειο της πόλης ε, και θα θέλαμε να εκφράσουμε τα συλληπιτεριά μας προς τις οικογένειες και επιθυμούμε να καταδικάσουμε αυτή την τρομοκρατική ενέργεια. Σήμερα εορτάζουμε την 60η επέτειο από την απόφαση του Στάλιν που οδήγησε στον θάνατο χιλιάδων αξιωματικών Πολωνών μετά από την εισβολή της Ρωσίας στην Πολωνία τον Σεπτέμβριο του 1939. Στην προηγούμενη θητεία μας ε, είχαμε την ευκαιρία στο Κοινοβούλιο να ε, δούμε μια ταινία που ήταν αφιερωμένη σε αυτό το επεισόδιο, το Κατίν. Αυτή η ταινία για πρώτη φορά προημερών ε, πέρασε και από την ρωσική τηλεόραση. Στις, σαν σήμερα το Κατίν, στην 7η Απριλίου, παρουσία του, του Προέδρου της ε, Ρωσίας αλλά και του Πρωθυπουργού της Ρωσίας εορτάζεται αυτή η επέτειος στην πόλη Κατίν. Πρόκειται για ένα μήνυμα το οποίο αποστέλλεται και σε ολόκληρη την Ευρώπη για το ότι το ανατολικό και δυτικό τμήμα της Ευρώπης βρίσκονται στην οδό της συμφιλίωσης, κάτι το οποίο υποστηρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια. Θα ήθελα να σας ενημερώσω επίσης ε, πως ε, κατά διάρκεια της ε, σημερινής μας συνεδρίασης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εκπροσωπηθεί από τον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς, τον Πρόεδρο Μπαρόζο για οικογενειακούς λόγους σημαντικούς. Δυστυχώς δεν μπορεί να παραστεί ανάμεσά μας σήμερα. Τα πρακτικά της συνεδριά ολομέλειας 25 Μαρτίου και όλες τις ε, αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου είναι στην διάθεσή σας. Έχετε παρατηρήσεις. εντάσεις, όχι, άρα μπορούν να εγκρινθούν τα πρακτικά. Ο κύριος Σπερώνη ζήτησε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εσείς ε, αναφέρατε τα θύματα της ε, τρομοκρατικής δράσης στην ε, Ρωσία, αλλά τρομοκρατικές ενέργειες έγιναν στο Αφγανιστάν, το Πακιστάν, το Ιράκ και αυτές είναι χώρες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ως εκ τούτου θεωρώ πως θα ήταν πρέπον να μνημονεύσουμε και τα θύματα αυτά. Έχετε δίκιο κύριε Σπερώνη.